good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ε, συνεδρίαση, να περάσουμε και στις ψηφορίες. Έχουμε πολλές ψηφορίες, ελπίσουμε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε μέσα στην επόμενη μια μισή ώρα. Σημείο 1, έγκριση της ημερησίας διάταξης. Έχω ένα σχόλιο κατόπιν αιτήματος ε, του εισηγητή Τη γνωμοδότηση ε, τη ΣΥΝΤΑ για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ και τη Συμφωνία Προστασία των Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ, που υποστηρίζεται από του και συζητητέ, προτείνω τι ακόλουθε αλλαγέ. Ε, οι ψηφοφορίε για τα σημεία 7 και 9 δεν θα λάβουν χώρα. Το σημείο 10 την Σύναψη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών ε, θα ψηφιστεί πρώτα και θα ακολουθηθεί από το σημείο 8 το μόνο μοθετικό συνοδευτικό ψήφισμα για την APA Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Αν συμφωνείτε, υιοθετείτε η ημερησία διάταξη με τις τροποποιήσεις που σας προανέφερα. Περνάμε στο σημείο 2. Αν Ανακοίνωση του Πρόεδρου δεν έχω ανακοινώσει. Σημείο 3. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου και 14 Οκτωβρίου. Έχετε σχόλια. Όχι από ό,τι φαίνεται. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο σημείο 4, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες σας έτοιμες. Η πρώτη ψηφοφορία αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον πλανήτη και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, της η έκθεση 2018. Θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια, την κυρία Βιζλερλίμα, αν θέλει το λόγο. Μια στιγμή. Υπάρχει πάρα πολύ θόρυβο στην αίθουσα. Μπορείτε να καθίσετε, παρακαλώ, ησύχως. Παρακαλώ. Δύο φορές έχουμε παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Θέλω σήμερα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συμμετείχαν ε, σε αυτές τις εργασίες, το προσωπικό, τους βουλευτές και να ευχαριστήσω και το κλίμα, το πολύ θετικό κλίμα μέσα στο οποίο έλαβαν χώρα συζητήσει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Ας περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Λοιπόν, χρειάζομαι την ένδειξή σου, Ρόκο γιατί έχουμε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Συμβιβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 226 τροπολογία υπέρ. Κατά. εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. εποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά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 Και πάμε στα εκτιμώντα. τροπολογία 57, υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 46, υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 68, urban Κρέσπο, υπέρ, κατά, Αποχέ. Να ελέγξουμε για την τροπολογία 68. Άρχεται η ψηφοφορία.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 απορριπτεται Απορρίπτεται. 35-29. Τροπολογίες 3 και 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές. Να αλλάξουμε το 5, τροπολογία 5 του κυρίου Ρούισεν. Λήξη. So, this amendment... Απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Και πάμε τώρα στις τροπολογίες 6, 7, 8 και 9, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 10, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 καταπίπτει. 12 και 13 καταπίπτουν 14, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε την 16. Ελεύθερη ψηφοφορία. Ελέγχουμε την 16 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 και 20 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε τη 19 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε τις 19 και 20 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτονται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Συγγνώμη, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 και 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόκειται εδώ για υπόψη. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 29. Άρχεται ψηφοφορία. Κάποιος λείπει. Λήξη. Εγκρίνεται. 30. 39,27 ήταν το αποτέλεσμα. 30 και 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται. 34 και 35 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτονται. 36 υπέρ εποχές, αποχές απορρίπτονται. 37-38 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτονται. 39 υπέρ κατά εποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 και 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 43 και 44 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε τις 43 και 44 άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτονται. Πάμε στη 45. Φαντάλερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 μέχρι 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51-52 υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται. 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Και φτάνουμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τρεις συνάδελφοι λείπουν. Ξυπνήστε. Τρεις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Λήξη. Εγκαταλείπω. Εγκρίνεται 48 υπέρ, 6 κατά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. We immediately move on to item number Περνάμε μέσα στο σημείο 5.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 Πάμε στην 125. Εξαιρετική προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 135 και αποσυρθεί, συμβαστική 11 υπέρ κατά. Εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν ψηφίζουμε την 192 τροπολογία του κ. Μπασέσκου υπέρ. Κατά. εποχές. Να ελέγξουμε την 192 άρχιτη ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 195 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. 195 έρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Μάλιστα, ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Πάμε στην 196 περ, κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω το απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε. Λήξη. Απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Αλλά να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά εποχές. Απορρίπτεται. 2.15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 2.22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 2.43. Κύριος και πέρα Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Συμβαστή 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, Συμβαστή 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, κατόπιν έχουμε την τροπολογία 289 του κ. Μπασέσκου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 290 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος, μάλιστα. Τη 290 άρχεται η ψηφοφορία. It's closed. Perhaps you have to have a look at the whole committee, not just... Uh, λοιπόν, προσπαθούμε να δούμε όλη την Επιτροπή. 2,91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2,92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2,93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 294 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 295 υπέρ κατά αποχές 2.95 D95 εγκρίθηκε, επομένως έχουμε αυτή την προσθήκη του κ. Καστάλντο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2,97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3,18 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 6. Εγκρίνεται. 319 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και πάλι την 319. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Λήξη. Απορρίπτεται. 320 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 322 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 324 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστή 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστή 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 333 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 334 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 335 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 356. Χαλίτσκι και Σικόσκι. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 357 Λόπες υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 358 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβεστική 36 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 372 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται, 373 υπέρ, κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 37 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται, 39 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 394 υπέρ, κατά εποχές να ελέγξουμε την 394, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Μάλιστα, ξεκάθαρο. 395 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 κυρία Πύρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 Ντάνσον υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 28, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη, εγκρίνεται. Συμβαστική 44, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 45, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 57 η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Η 57. Πάμε στα υπόψη. 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ερπολογία 7 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και μπορούμε να περάσουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία του συνόλου της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε έρχεται η ψηφοφορία Τέσσερις λείπουν. Τρεις, δύο, ένας. Όλοι ψήφισαν, λήξη. Εγκρίνεται 47 υπέρ 12 κατά. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε. Να ευχαριστήσουμε τους κοιόδης εισηγητές, ήταν έξοχη η συνεργασία. Πάμε στο σημείο 6 εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ετήσια έκθεση 2018 και ως Ντανζόν εισηγητής θέλει να πάρει το λόγο. Ουχή. Εν τη αυτή περιπτώσει ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Συμβαστική ένα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, καταπίπτουν όλα αυτά. 47. Η 39 δεν εγκρίθηκε, οπότε πάμε 42, κυρία Νόημαν. Υπέρ της κυρίας Νόημαν, της τροπολογίας κυρίας Νόημαν. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 82 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95. Πάει και άλλος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 97. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 101 καταπίπτει. Απορρίφθηκε η 100. Η 101 καταπίπτει αν εγκριθεί η 100. Α, τι κάτι μου λείπε, κάτι μου λείπε, εντάξει. Η μεγάλη στιγμή του Μιχαήλ Γκάλερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 102 καταπίπτει. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. οκτω συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119-120 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτωτε. 136 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 142, 143 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ να ελέγξουμε 145 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Τι 148 εννοούσα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 152. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 149 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για την 150 του κυρίου Καστάλτο. Πέρας. Εγκρίνεται. 26-25. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε όμως. 153 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έλεγχος. Μου λένε ότι 153 καταπίπτει από ό,τι φαίνεται. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε. Εντάξει με την 153. 151. Πρέπει να ψηφίσουμε την 151. Ωραία. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 151. Άρχεται η ψηφοφορία. Έρας. Εγκρίνεται σαφώς. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 159 άρχεται. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Εκατόν Μιχαήλ Γκάλερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 160. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για την 164 άρχεται. Πέρας απορρίπτεται, ξεκάθαρο. 162 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 168 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 169, 170 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 171 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 172 καταπίπτει, καλά μαντάτα. Πάμε ήδη στην 181. Φοργόντας Μάνι, Μπάνιον, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 190, ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. 198. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 203 και 204 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος για τη 202 της κυρίας Κάνκο. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 202. Πέρας. Εγκρίνεται. 201. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Α, απορρίπτεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 207 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 212 της κ. Κανιέται υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 212 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.14 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για τη 214 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. 2.16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχος. Εντάξει. 2.16 της κυρίας Νόημαν. Πέρας. Απορρίπτονται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 229 ξεκινάει τώρα πέρας απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15, ναι. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.54 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 254 άρχεται πέρας εγκρίνεται λοιπόν 255 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 255 άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. «259 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». «257 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». «258 υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχος για τη 258, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 260 κατά πίπτη. πάμε 261 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 262 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 263 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 266 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για τη 266 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 265 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 265. Πέρας και νίκησε η κυρία Νόημαν. Δεν χρειάζεται να ελέγχουμε πλέον. Εγκρίθηκε η 265. Η 264 συνεπώς καταπίπτει. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2,75 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. κατά καταπίπτει. Τι θέλουν αυτοί εδώ πέρα. 2.83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.94 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη 2.94 άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. 2.95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για τη 2.97. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται ξεκάθαρα. 298, 299, 300 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 301 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. Την τροπολογία του κυρίου Καστάλντο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 302 του κυρίου Πέτρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 303 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 303 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 304 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 305 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 314 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 315-316 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 317 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 318 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 322 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 325 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 320 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 320. Ξεκινάει τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 324 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 324. Ξεκινάει τώρα. Εγκρίνεται. Τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 326 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε μια σελίδα. 340 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 340 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτωται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 347 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 348 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 349 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 350 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. 378. Τζέφρι Βανόρντεν και άλλοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 379 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 387. Σικόρσκι υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος για την 387. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 388 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την 388. Άρχεται η ψηφοφορία. 388. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 389 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε και την 389. Μήπως δεν έχω το σωστό κατάλογο ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. 390 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 391 ψήφι περ Κατά αποχές απορρίπτεται. 394 ψήφι περ κατά αποχές απορρίπτεται. 392 ψήφι περ κατά αποχές απορρίπτεται. 395 ψήφι περ κατά αποχές απορρίπτεται. 396 ψήφι κατά αποχές θα ελέξουμε την 396 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Βασιχώς και τώρα είναι η επόμενη αντιπρόεδρος. 393 ψήφι πέρα κατά αποχές. Θα ελέξουμε και αυτή την τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 405 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 406 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 407 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 408 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 409 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 410 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστικό 7 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 418, πάει και άλλοι. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 419 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 420 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 421 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 422 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 423 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε την 423 έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 424 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 432 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 427 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 425 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε την 425, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 431 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έχουμε τις ταυτόσιμες τροπολογίες 429-430 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 428 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, εντάξει. Ελέγχουμε την 428 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. η επόμενη. 4.33 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε την 4.33, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Πηγαίνουμε τώρα στην 437 πάει και άλλη ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 438 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 440 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 439 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 451 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε, εντάξει, την 451 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε, ήταν σαφές. 452 ψήφι υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε την 452. Πέρας απορρίφθηκε. 453 ψήφι πέρα. Συγγνώμη, πρόεδρος. Ξέχασα την 454 Νόημαν. Ψήφι ΠΕΡ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 453 ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 455 ψήφι πέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 457 ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 456 ψήφι κατά, αποχές εγκρίνεται. 4.58 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4.59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4.60 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4.61 ψήφι υπέρ. Συγγνώμη, λέω προς 4.64 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4.63 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 462 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε την 462. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε 31 προς 30. Κατά πίπτη 461. Πηγαίνουμε στην 466. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 467. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την 467. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 468 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 469 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 470 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 471 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 472 υπέρ, κατά, αποχές, Λέω να ελέγξουμε την 472 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται σαφώς. Συμβιβαστική 29 ψήφι ΠΕΡ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 482 Γλουξμάν και άλλοι ψήφι ΠΕΡ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, ναι. 482 αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, πράγματι, εγκρίθηκε. Είχατε δίκιο. 483 ψήφι πέρυ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία την 483. Πέρας. Απορρίφθηκε. 484 ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 485 ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 485 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 486 ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η Αύκο τι θέλει εδώ. Τέλος πάντων. Αύκο 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αύκο 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την Αύκο 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αύκο 7 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την Αύκο 7. Άρχεται η ψηφοφορία. It's closed. Πέρας. Απορρίφθηκε. ΑΦΚΟ 8. Ορίστε. 24 προς 37 ήταν το αποτέλεσμα. Αύκο 8. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 9. Ψήφι υπέρ. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την αύκο 8. Άρχεται η ψηφοφορία. closed. Rejected. Απορρίφθηκε. Αύκο 9. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αύκο 10. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω θα ελέγξουμε τη 10. Άρχεται η ψηφοφορία. closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αύκο 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αύκο 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αύκο 20 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε την 20 της Επιτροπής Γιατί ήταν αμφίροπο το αποτέλεσμα. Πέρας. Όχι, δεν ήταν. Απορρίφθηκε. 21 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 22 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε την ΑΦΚΟ 22, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Ρητολικές αναφορές 1 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, θέλετε να ελέγξουμε το citation 3, την ρητολογική αναφορά 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 47 προς 11. Εγκρίθηκε. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7. Υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε την 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε σαφώς 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 9 άρχεται ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία για την 12. Πέρασε απορρίφθηκε 30 προς 32 η ψήφη κατά ήταν 32 και φάσαμε στην τελική ψηφοφορία για την έκθεση όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε 41 ψήφη, πέρι 22 κατά δύο αποχές συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Μισό λεπτάκι, κύριε Γουόλας. Εκτός μικροφώνου. Ο κύριος Γουόλας εκτός μικροφώνου. Η ομάδα μας, NGL, θα καταθέσει έκθεση μειοψηφία ε, για αυτήν την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Γουόλας. Και τώρα πηγαίνουμε στις εκθέσεις για το Βιετνάμ. Από ό,τι με ενημερώνουν αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία του σημείου 8. Έτσι έχει κατάσταση. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο νέο. Ωραία. Έτσι θα προχωρήσουμε. Θα ψηφίσουμε καταρχάς για το σημείο 8. Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και τη Σοσιαλιστική Δημοκρατίας του Βιετνάμ αφετέρου. Η συγγήτρια, η συγκεκριμένα συντάκτρια γνωμοδότηση είναι η Ιζαμπέλ Βίζελερ Λίμα. Θέλετε το λόγο Ιζαμπέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο λέξεις στα γαλλικά. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και για το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε. Ποτέ δεν είναι εύκολο να ε, καταλήξουμε σε συμφωνία. Εδώ το καταφέραμε σε σχέση με το τι εμείς επιθυμούμε, πού θέλουμε να καταλήξουμε. Δηλαδή θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. και που δεν συμφωνήσαμε είναι ποιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθήσουμε για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Συμφωνούμε πάντως απόλυτα ως προς το ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο προορισμός μας. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να ψηφίσουμε επί του ψηφίσματος, χωρίς όμως να ψηφίσουμε ε, το consent, ε, γιατί έτσι αυτό τουλάχιστον αποφάνθηκαν ε, όσοι διαπραγματεύτηκαν, αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να στείλουμε ένα χειρό πολιτικό μήνυμα, διότι αν επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, το αποτέλεσμα θα είναι σχεδόν ομόφωνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, γιατί όλοι δείξατε προσήλωση, αφοσίωση, ώστε ως Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να στείλουμε ένα πάρα πολύ χειρό μήνυμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο, όχι, επομένως. Προχωρούμε. Με βάση τον κατάλογο. Η τροπολογία 1 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Καταπίπτει οι δύο. Δεν θα ψηφίσουμε την τροπολογία 4. Πηγαίνουμε στη συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 δεν ψηφίζουμε. Συμβεβαστική 3 ψήφι περ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στο τροπολή 22 χάουταλα ψήφι περ, κατά αποχές. Ορίστε. Όχι. Ψηφίσαμε την τροπολογία τη συμβιβαστική 4 και είμαστε στην 22. Ψήφι υπέρ, κατά, εποχέ. Θα ελέγξουμε την 22. Μετά είναι 20, συγγνώμη, συμβιβαστική 5. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 22. Πέρας. Απορρίφθηκε. Και τώρα ερχόμαστε στη συμβαστική 5. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. It's closed. ψηφοφορίας εγκρίνεται ξεκάθαρα και ήδη φτάσαμε Ήδη φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότης όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία. Λείπουν δύο. Πέρασε εγκρίθηκε 48 υπέρ, 8 κατά, 6 αποχές. Και τώρα πηγαίνουμε στο σημείο 10. Αυτή η λίστα, έτσι, ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνία έφεση των αλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ. Συμβιβαστική 1 ψήφι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία. πέρας Εγκρίθηκε. Συμβαστική 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά, ονομαστικά, ψηφίζουμε, άρχεται. 5, 4 λείπουν, 3 λείπουν, 2. 2. Πέρας ψηφοφορίας. 47 υπέρ, 7 κατά, 8 αποχές. Και με αυτά και με αυτά περάσαμε μια μισή ώρα ψηφοφορίες. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, που ήταν εδώ και ευθύ αμέσω προχωρούμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Παραμένουν ε, όσοι πρέπει να είναι εδώ, οι υπόλοιποι να περάσουν τώρα και θα τα πούμε το μεσημέρι.